θέση του από την 4η Ιανουαρίου 2012. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία και σύμφωνα με το άρθρο 74 του εσωτερικού κανονισμού θα υπογράψουμε μία πράξη η οποία θα, της οποίας ο τίτλος βρίσκεται εις ε, τα πρακτικά. Και ερχόμαστε τώρα εις ε, την τελική ημερήσια διάταξη, το τελικό σχέδιο της ημερησίας διατάξεως και ε, έχετε το, το τελικό, τελική μερίσια διάταξη την οποία υιοθέτησαν οι, οι πρόεδροι των επιτροπών που έχουμε διαπραγματευτεί με τις διάφορες πολιτικές ομάδες κατόπιν διαβουλεύσεων και με τη στήριξη όλων των πολιτικών ε, ομάδων θέλω να σας παρουσιάσω τις τελικές αλλαγές. Ε, τετάρτη Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, δύο εκθέσεις του κυρίου ο ΡΑΠΚΑΙ καταρχήν η αίτηση υπεράσπισης της ατσιλίας και των προνομίων του κυρίου Σπατσικίτς που θα συζητηθούν και τα δύο σημεία από κοινού και αυτά μόλις ολοκληρωθεί η οθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση. Την... Ε, την οποία υιοθέτησαν οι πολιτικές ομάδες. Μετά, σχετικά με την προφορική ερώτηση που απευθύνεται εις το το Συμβούλιο. Ο κύριος ε, Ραπκάη έχει μία έκθεση σχετικά με την ασυλία του κυρίου Ντεμαγκίστριξ που επίσης θα συζητηθεί και ε, γι' αυτό έχουμε μεταφέρει αύριο τις ψηφοφορίες στις 14.00 και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι στις 12. Αυτές είναι οι οι παρατηρήσεις οι δικές μου. Αν εσείς δεν έχετε παρατηρήσεις ε, σχετικά ε, με ε, τις αλλαγές της μελητησίας διατάσεως, υιοθετούνται. Τώρα έχουμε ε, την ε, ε, ημερήσια διάταξη και μπορούμε αμέσως να προχωρήσουμε στην εξέταση της ημερησίας διατάξεως διότι όπως γνωρίζετε το πρώτο σημείο αλλά βλέπω ο κύριος Βαντάλεν θέλει κάτι να πει. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να αντιδράσω στις ανακοινώσεις που κάνατε όσον αφορά την Αίγυπτο. Εγώ ήμουν στο Κάιρο στις εκλογές μαζί με αντιπροσώπους του Ινστιτούτου Κάρτο που ήταν καλεσμένοι για να ελέγξουν τις εκλογές. Είδανε, διαπίστωσαν κάποιες, ε, ε, κάποια πράγματα τα οποία δεν πήγανε καλά και θα ήθελα κι εγώ να τα αναφέρω αυτά για να τα έχει υπόψη της Ερμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να τα ξέρει και να ενημερώσει σχετικά και τις Αιγυπτιακέ ε, Αρχές. Θα σας στείλω γραπτά ό,τι παρατηρήσει έχω να κάνω. Ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση. Μπορώ να σας πω ότι ευχαρίστως ε, δεχόμαστε τις παρατηρήσεις και σημειώνουμε αυτά τα οποία είπατε και δίνω το λόγο στον κύριο Ντόλ. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλό. Αύριο στις 2 η ώρα είπατε για την ψηφοφορία αυτό, είπατε. Όχι. Όχι, μπορεί να τραβήξει ως τις δύο. Δηλαδή οι ψηφοφορίες μπορεί να τραβήξουν ως τις δύο. Όχι θα ξεκινήσουν στις δύο διότι θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς και όλες τις επεξηγήσεις ψήφου. Δεν πρόκειται μόνο για τις ψηφοφορίες, αλλά όλες τις επεξηγήσεις ε, ψήφους που συνήθως μπορούν να κρατήσουν έστω και μία ώρα. Ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί και να ε, μπορέσει να εκφραστεί κατά τις επεξηγήσεις ψήφου. Ο κύριος Ντεσιλβέστρης ε, διαδικαστικό. Όπως και ο κύριος Ντόλ, ομολογουμένως δεν κατάλαβα και εγώ καλά περί την πρόκειται. Θα συζητήσουμε για το αίτημα της ασυλίας του κυρίου Ντεματζίστρης που ούτε καν είναι πλέον ε, συνάδελφός μας. Δεν είναι πλέον βουλευτής. Αυτό θα συζητήσουμε αύριο γιατί δεν καταλαβαίνω. Ε, ε, αξιότιμε κύριε αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό διότι είναι ένα καθήκον που έχουμε αναλάβει και σύμφωνα με, την με τον εσωτερικό κανονισμό έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ο κύριος Πόσελ τώρα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά αύριο έχουμε μία από τις πλέον βασικές ψηφοφορίες αυτής της θητείας, δηλαδή η σύνομη ψηφοφορία για την προσχώρηση της Κροατίας, για την οποία χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία θα παρακαλούσα λοιπόν να τοποθετηθεί αυτή η ψηφοφορία στην αρχή για να μπορέσουμε να έχουμε ε, ενισχυμένη πλειοψηφία. Είναι μία από τις πλέον βασικές ψηφοφορίες της ε, θητείας αυτής. Ε, θέλω... Συνάδελφοι, στις 12 θα ψηφίσουμε, δεν αλλάζει αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και μία από τις πρώτες ψηφοφορίες. Ε, σήμερα θα συζητήσουμε για την ε, Κροατία, για τη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας. Σήμερα συζήτηση, αύριο ψηφοφορία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Όντω, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ούτω ώστε να έχουμε την ειδική πλειοψηφία ε, στι ψηφοφορίε, το μέτρο που συμφωνούμε, εξυπακούεται. Ε, υπάρχει άλλη ερώτηση, βλέπω, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας. Ε, σας ευχαριστώ που θα ε, εξακριβώσετε τι γίνεται αύριο και αν αυτό συνέβη με τον ιστορικό κανονισμό. Ευχαριστώ που δείχνετε κατανόηση. Λοιπόν, η συζήτηση που θα γίνει αύριο για την άσκηση της ασυλίας του κυρίου Ντεματζίστρης είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε δράση. Ε, θα ήθελα δηλαδή να έχω την ευκαιρία να παρέμβω και στη συζήτηση. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι στα πλαίσια της διαδικασίας ε, ή Δεν θέλω να συμπιέζουμε έτσι τους κανονισμούς. Ε, θέλω να προβλέψουμε μέσα στον κανονισμό ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος ε, για το ΚΑΤΣΙΑ για να μπορέσουμε να παρεύουμε αν θέλουμε. Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να φοβάστε ότι δεν πρόκειται να σεβαστούμε τον εσωτερικό κανονισμό. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μία άσκηση εκενώσεως του κτηρίου. Παρακαλώ να εξέλθετε αμέσως και να φύγετε από το κτίριο όπως θα σας οδηγήσουν οι δυνάμεις ασφαλείας ε, και θα ειδοποιηθείτε όταν θα συνέλθει και πάλι η Ολομέλεια. Mrs. Sarizlowski. Hamburg-Erzburg-Delta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 Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι. Ήταν μια άσκηση μόνο αυτή, εκένωσης κτηρίου.